Καθίστε παρακαλώ. ναι, ναι, ξέρω. Κυρίε και κύριοι, έχει γίνει ένα λάθος στο λογισμικό και δεν έχετε τα συνήθη ονόματα στην θέση σας. Μπορεί να δείχνει ένα άλλο όνομα. Αλλά προσπαθούμε να το διορθώσουμε το συντομότερο δυνατόν. Αλλά επειδή θέσεις υπάρχουν άφθονες, αν δεν θέλετε να καθίσετε σε θέση που δεν γράφει το όνομά σας και ψάχνετε πού αναγράφετε το όνομά σας, σας παρακαλώ να το κάνετε αργότερα. Κύριος Μαριάς. Πρόεδρε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο που αναγράφονται οι θέσει. εγώ έχω βάλει την κάρτα μου αυτή τη στιγμή και παρά τα αυτά αναγράφεται το όνομα ενός άλλου συναδέλφου. άρα είναι θέμα ότι ακόμη και την κάρτα να βάλουμε που μπορούμε να τη βάλουμε σε όποια θέση δεν φαίνεται το όνομά μας αλλά υπάρχει εκεί πρόβλημα όσον αφορά την ψηφοφορία.